πιο πολλοί δουλεύουν στις μέρες μας ε, στη δημιουργία δημιουργικού παρά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Εδώ λοιπόν μιλάμε για την πολιτισμική πολυμορφία, για τον πλουραλισμό. Η οδηγία υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να δείξουν σεβασμό προς τους δημοσιογράφους, προς τους δημιουργούς, παρέχοντας και νομική ασφάλεια, η οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Εγγυάται δικαιώματα και ευνοεί την πρόσβαση στη γνώση, προάγει τα δικαιώματα των δημιουργών, προστατεύει τους δημιουργούς. Αυτό ακριβώς προστατεύουμε και εμείς τη δημιουργία ε, εκ μέρους των δημιουργών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτεκ για ένα λεπτό. Αυτή η εκδοχή της οδηγίας εισαγάγει λογοκρισία, ένα επίπεδο λογοκρισίας που δεν είχαμε στις πρώην κομμουνιστικές χώρες. Δείτε τι λέει το κείμενο το ίδιο. Δεν μπορείτε να πείσετε τα μέλη εδώ όλοι έχουν οχυρωθεί πίσω από τις θέσεις τους ε, πολίτες της Ευρώπης. Εάν δεν θέλετε να χάσετε τις ελευθερίες σας, τότε θα πρέπει να πείσετε τις κυβερνήσεις σας ίσως να ε, αποχωρήσουν. Θα έπρεπε να πείσετε τις κυβερνήσεις σας να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε, ας εγκαταλείψουμε αυτό το γραφειοκρατικό τέρας που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας δημιουργήσουμε μία πραγματική ένωση των εθνών. Μία καινοτόμα ένωση των εθνών. Τι σας σταματάει από την καταψήφιση αυτού του κειμένου. Υπάρχει μία μπλε κάρτα. Θα δεχτείτε την μπλε κάρτα του κυρίου Στρογεύσκη. Δέχεστε την ερώτηση του κυρίου Στρογεύσκη. Τη Σας ευχαριστώ πολύ. Είπατε κύριε ότι ε, αντιτίθεστε σε αυτή την οδηγία, άρα να μην αμείβονται οι ε, δημιουργεί. Εσείς ε, είσαστε υπέρ ενός κόμματος που στοχεύει στην αποχώρηση έτσι ώστε η χώρα μας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και άλλη ε, μπλε κάρτα. Ο κύριος Καβαντά. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα ο συνάδελφος ο οποίος ε, μας πείθει, θέλει να μας πείσει να αποχωρήσει από την να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε γιατί αυτός παρίσταται εδώ όταν του δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Μικρόφωνο. Απάντηση με μικρόφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Ναι, βεβαίως έρχομαι εδώ και ε, ε, δημοσία τάσομαι υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θεωρώ ότι και άλλες χώρες θα πρέπει να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σχηματίσουν μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση όχι ε, αυτό το γραφειοκρατικό τέρας, να δημιουργηθεί μία νέα Ευρωπαϊκή Ένωση καινοτόμα. Αυτό θα ήθελα να επισυμβεί για την Πολωνία ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θεωρώ ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάξει στάση, τότε θα πρέπει να αποχωρήσουμε και αυτό αφορά και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν περάσει πολλοί νόμοι και νομοθεσίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η θέση μου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, απαντήσατε σε μία ερώτηση από τις δύο, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω άλλο χρόνο. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Σαλίνη. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Άξελ Βός για την εξαιρετική του εργασία μέχρι τούδε. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες μάχες της τρέχουσας θητείας, γιατί Ευρώπη σημαίνει δημιουργία, εργασία και τέχνη. Πρόκειται για μία μάχη υπέρ της Ευρώπης. Ακριβώς για τι προασπίζομαστε αυτές τις αξίες. Αυτοί που καταφέρονται κατά της οδηγίες θα πρέπει να δουν τι κάνουν οι πλατφόρμες. Εάν θέλουν να εισπράξουν δις δολάρια, θα πρέπει τότε να αναγνωρίσουν την εργασία του δημιουργού που τους επιτρέπει αυτά τα έσοδα. Δηλαδή στο Google να υπάρχει Φυσικά να υπάρχουν διαφημίσεις, αλλά να αμείβονται οι δημιουργοί. Ε, κύριε Ρέντα, μιλήσατε για νέους. Υπάρχουν νέοι που πληρώνονται 3 ευρώ το κομμάτι για την εξαιρετική τους δημοσιογραφία. Εάν θέλετε να τους υπερασπιστείτε, να υπερασπιστείτε το copyright. Για ένα λεπτό ο κύριος Γραμματικάκης έχει το λόγο η μάχη για τα πνευματικά δικαιώματα ξεκίνησε ως μια τεχνική συζήτηση στην πορεία όμως εξελίχθηκε σε μάχη για την ψυχή της ευρώπης δηλαδή τον πολιτισμό και τις αξίες της. η συμφωνία δεν εξασφαλίζει μόνο ότι οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί θα επιβιώσουν στην ψηφιακή εποχή αποδεικνύει επίσης κάτι σοβαρότερο ότι η ευρωπαϊκή ένωση έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει τους τεχνολογικούς κολοσσούς και τις δυνατότητές τους να παραπλανούν πολίτες και πολιτικούς και εντυπωσιάζομαι από το ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν αυτό. μετά από δυόμιση χρόνια διαπραγματεύσεων λοιπόν και τρεις διαφορετικές επιτροπές πέντε και τρεις ψηφοφορίες στην ολομέλεια έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η οδηγία υποστηρίζεται από όλους τους επίσημους φορείς που πολύ την έχουν συζητήσει δημιουργών και καλλιτεχνών. Ως συζητητής του Σοσιαλιστών στην Επιτροπή Πολιτισμού θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω όλους τους συναδέλφους που τάσσονται υπέρ του ανοιχτού και ελεύθερου διαδικτύου και δίκαιου όμως διαδικτύου να στηρίξουν το αποτέλεσμα του τριλόγου. Δεν θα είναι μια μάχη μόνο για το παρόν της Ευρώπης αλλά επίσης αγαπητοί συνάδελφοι και για το μέλλον της. Ένα λεπτό κύριο Σούλικ. Ευχαριστώ πολύ. Η οδηγία, η τρέχουσα οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα θα ε, αλλάξει επιταχύρω, ιδίω ό,τι αφορά το άρθρο 13 με την νέα αυτή πρόταση και το ίδιο θα γίνει και με το άρθρο 11. Ουσιαστικά θα περιλαμβάνονται και τα πολύ μικρά αυτά αποσπάσματα, παραθέματα που δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο τι σημαίνει αυτό. Κοινωνικές πλατφόρμες είναι αυτές που θα εξασφαλίζουν ε, την αποτροπή κλοπής περιεχομένου Δηλαδή αυτός που έχει ένα χώρο στάθμευσης, πάρκινγκ, θα είναι υπεύθυνο για το ενδεχόμενο κλοπής ε, κάποιου αυτοκινήτου ή απώλειας αντικειμένου μέσα από το αυτοκίνητο. Εκπλήσωμε επίσης ε, που δεν λαμβάνει υπόψη τη την κοινή γνώμη Κομισιόνα. Για τάρτα 11 και 13 έχω υποβάλει ε, τροπολογίες διαγραφής. Ευχαριστώ. Μπόγκοβιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Όλοι έχουμε το δικαίωμα ε, της ελευθερίας έκφρασης. Μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα στο διαδίκτυο, αλλά έχουμε και το δικαίωμα ε, της προστασίας. Θέλουμε ψηφιακό περιεχόμενο, ε, θέλουμε πνευματικά δικαιώματα, θέλουμε ελευθεροτυπία. Αλλά Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των δύο κατηγοριών δικαιωμάτων. Αυτό δεν ισχύει. Ο Άξελ Φώσε κάνει πολύ καλή δουλειά. Εστιάζουμε ουσιαστικά στις ε, μεγαλύτερους κολοσσούς ε, του διαδικτύου, πλατφόρμες που αποκομίζουν ε, τεράστιο κέρδος, αλλά δεν μοιράζονται το κέρδος αυτό με τους δημιουργούς. Αν θέλουμε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, και ανεξάρτητους ε, δημιουργούς γενικώ και καλλιτέχνες θα πρέπει να την εγκρίνουμε την πρόταση αυτή. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τους μεγάλους αυτούς ε, ομίλους, ε, αλλά θα προστατεύσουμε τη δημιουργία. Θα στηρίξω λοιπόν την έκθεση αυτή, γιατί θα προωθεί την ισότητα. Ευχαριστώ κύριος Μπλάνκο Λόπεθ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κανένας δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ανελευθερία στο διαδίκτυο, γιατί το διαδίκτυο δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς νόμους, αλλά δημιουργία υπάρχει μόνο αν υπάρχει δίκαιη αμοιβή. Αυτή η οδηγία προσπαθεί να διορθώσει αυτές τις ανισορροπίες για να ενισχύσει τους δημιουργούς, να δώσει χώρο στη αλυσίδα αξιών. Δεν καταλαβαίνω πώς ε, πολλοί εκπρόσωποι της αριστεράς δεν δέχονται τον πλούτο των πλατφορμών λέγοντας ότι υπερασπίζονται τους δημιουργούς. Δεν υπάρχουν ούτε μέμ ούτε hyperlinks. Αυτό αυτό είναι το διαδίκτυο του 21ου αιώνα. Είναι η ελευθερία του εκφράζεστε, η ελευθερία δημιουργίας και η σωστή αμοιβή των δημιουργών. Κύριε Μπλάνκο Λόπεθ, έχετε δύο μπλε κάρτες. Τις δέχεστε? Ο κύριος Ρούμπιχ και η κυρία Ματίας θα υποβάλουν την ερώτησή τους σε 32. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπλάνκο Λόπεθ κατά πόσον ισχύει ότι στο μέλλον ε, όταν κάποιοι αναφορτώνουν δεν θα έχουν ευθύνη όλοι ουσιαστικά όσοι δεν είναι επιχειρηματικοί. Κυρία Ματίας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συναδελφό που είπε ότι δεν υπάρχει δημιουργία, αν δεν υπάρχει σωστή αμοιβή, θα ήθελα να διαβάσει την οδηγία εκεί που λέγεται ότι θα υπάρχει δίκαιη αμοιβή για τους ε, δημιουργούς. Εγώ δεν το βλέπω πουθενά αυτού. Πείτε μου πού αναφέρεται η δίκαιη αμοιβή για τους δημιουργούς. Βρείτε μου το παράθεμα. Μη λέτε λόγια θα πρέπει να επανισορροπήσουμε την αλυσίδα αξιών. Οι πλατφόρμες συνεισφέρουν για την δίκαιη αμοιβή, δηλαδή ανταμείβεται η εργασία, η δημιουργία δεν την χάνει εκμετάλλευσης. Δεν καταλαβαίνω γιατί η αριστερά θέλει να ευεργετούνται μόνο λίγοι ε, σε σχέση με τους δημιουργούς της Ευρώπης μας, των χωρών μας. Δεν είμαι σίγουρη ότι απαντήσατε στον κύριο Ρούμπιχ. Κύριε Μπλάνκο Λόπεθ, σας ε, υπέβαλε ερώτηση και ο κύριος Ρούμπιχ. Δεν απαντήσατε. Υπέβαλε την ερώτηση. Θυμόσαστε τι σας ρώτησε ο κύριος Ρούμπιχ. Κύριε Ρούμπιχ, μπορείτε να επαναλάβετε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπλάνκο Λόπεθ κατά πόσον ισχύει ότι οι χρήστε μα επαγγελματικοί δεν έχουν πλέον ε, κάποια ευθύνη ε, και ε, επομένω δεν μπορούν να, να, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια προσβολή για την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία για το περιεχόμενο το οποίο βρίσκεται σε κάποια πλατφόρμα από απλού χρήστε. Δεν είναι επαγγελματικοί. Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένο το κείμενο που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα όλων των μερών. Για τον αθλητισμό όμω, το ότι δεν συμπεριελήφθη δική μνήμα στα δικαιώματα των διοργανωτών αθλητικών διοργανώσεων είναι κακό. Είχαμε το τροπολογία στο αρχικό άρθρο 12. 400 ψήφισαν υπέρ την προηγούμενη Ολομέλη του Σεπτεμβρίου για αυτό το θέμα. Θα θέλαμε να είχε υπάρξει μια τολική σκέψη ε, για την απόφαση Premier League Marfin ε, που σημαίνει θα μπορούσαν να υπάρχει αυτή η προστασία των αθλητικών διοργανώσεων από τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν θα ανέλυε τα σχετικά συστήματα προστασία. Τελικά η επιλογή είναι μόνο μια γενική δήλωση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα των δημιουργών αλλά και των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων. Επομένως, ε, θα ψηφίσω το κείμενο, ε, γιατί παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προστατεύσουν τα δικαιώματα των δημιουργών, αν και θα ήθελα και κάτι παραπάνω για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων. Ευχαριστώ κυρία Ρέγνερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση εδώ ε, δείχνει ε, πόσο πάθος ε, μας χαρακτηρίζει στον κοινοβουλευτικό μας βίο. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας, αλλά σίγουρα δεν βαρεθήκαμε σε αυτή τη συζήτηση. Τα δικαιώματα των πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να προσαρμοστούν στην σύγχρονη πραγματικότητα. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν κερδίζουν πάρα πολλά, που δεν γράφουν το best seller και έχουν ε, λογαριασμούς ε, εκατομμυρίων. Για αυτούς η ε, κατάσταση γίνεται όλο και πιο επισφαλής και ιδίω ό,τι αφορά τα πνευματικά του δικαιώματα. Εμείς θέλουμε όχι να καταστρέψουμε το ελεύθερο διδίκτυο, αλλά να προστατεύσουμε τα δικαιώματα. Θέλουμε επίσης όλοι να, να προστατεύσουμε την ελευθερία έκφρασης για όλους, αλλά θέλουμε ε, και την προστασία των δημιουργών. Θέλουμε ευθύνη για τις ε, πλατφόρμες. Αυτό οδηγεί όμως σε φιλτραρίσματα, ε, στο upload filters. Εγώ θεωρώ ότι σε όλο αυτό είναι η σημασία η κεντρική που έπρεπε να έχει προστασία των δημιουργών. Άρα πρέπει να υπάρχει δίκαιη αναλογική αμοιβή για τους δημιουργούς. Γι' αυτό δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη για το αποτέλεσμα της προφορίας στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Μπαίνουμε στη διαδικασία. Κάτσε Η πρώτη ομιλήτρια, η κυρία Σόιτρόβα. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Άξελ Φως, τον εισηγητή για την ευσυνείδητη εργασία του και το γεγονός ότι ήταν πολύ θαραλέος γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μία μεγάλη εκστρατεία. Ε, Πιστεύω λοιπόν ότι έχει φτάσει σε μια εξισορρόπηση μεταξύ πλατφορμών, δημιουργών και ημών των χρηστών. Οι μη εμπορικές πλατφόρμες όπως ο Wikipedia και άλλες έχουν γίνει αποδεκτές και το άρθρο 13 τάσεται κατά της λογοκρισίας. Αυτοί που αντιτίθενται δεν προβάλλουν μία ε, επιχειρηματολογία. Πώς όμως θα αμείβονται σωστά οι δημιουργοί αν δεν υπάρχει το άρθρο 13. Εμείς θα πρέπει να έχουμε πολύ ε, καλής ποιότητας ε, έργαση. Η κυρία Κονέτσνα προβάλλει μία μπλε κάρτα και δεν προβλέπεται στη διαδικασία Catch the Eye. Κυρία Σόιντροβα, την δέχεστε? Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σόιντροβα εάν μιλά για μια συντονισμένη καμπάνια τι εννοεί όταν μιλά για εκδότες, εκδότες που απειλούν τους δημοσιογράφους και στην περίπτωση αυτή θα υπάρξουν συνέπειες, δηλαδή αν υπάρχει έλεγχος περιεχομένου. Τι εννοείται, πρόκειται για μία ποταπή συναλλαγή, τίποτα άλλο. Απλώς έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Κυρία Σόιντροβα, θα ήθελα να πω ότι ότι ε, εκτιμώ σε αυτή τη συζήτηση τις ε, δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, το ανοιχτό πνεύμα και τη διάβια. Αν εσάς μπορούν να σας εκβιάσουν, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Εγώ δεν υφίσταται κανέναν εκβιασμό. Πρέπει να βρούμε μια δίκαιη λύση για όλους τους δημιουργούς. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε δεχόμαστε κακόβουλους χειρισμούς. γυλάρια ένα λεπτό μετά από τρία χρόνια εργασίας θα πρέπει να φτάσουμε σε μια λύση που να είναι δίκαιη και εξισορροπημένη. Αλλά δεν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα όμως και η ελευθερία του εκφράζεστε, η καλλιτεχνική δημιουργία, το έρευνα. Αυτό λέει το Σύνταγμά μας, αλλά και η Χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και φυσικά η αλυσίδα αξιών είναι η δημιουργή έναντι των γιγάντων του διαδικτύου που χρησιμοποιούν τα δεδομένα και δεν καταβάλουν φόρους, χρησιμοποιούν τρόλ έτσι ώστε να εξοριγνύουν στοιχεία. Μετά από αυτή την οδηγία, θα υπάρχει όμως το διαδίκτυο, αλλά και η ελευθερία του εκφράζεστε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρίνιο Ιππίντο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, εγώ κατανοώ τη θέση των GAFA, Google, ε, Apple, Facebook και Amazon που όλοι αντιτίθενται σε αυτή την οδηγία γιατί απειλεί τα δυσθεώρητα κέρδη στα οποία έχουν φτάσει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή προστατεύεται το περιεχόμενο των δημιουργών, εκδοτών και συγγραφέων. Καταλαβαίνω γιατί η γκάφα αντιτίθενται σε αυτό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κόμματα πειρατών, κόμματα κατά της δημιουργίας και των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Και καταλαβαίνω γιατί και η άκρα δεξιά αντιτίθενται σε αυτά τα ε, πνευματικά δικαιώματα. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε την, τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Καταλαβαίνω γιατί η άκρα δεξιά αντιτίθεται. Πιμέντο Λόπες. Ευχαριστώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα συμφέροντα των γιγαντιαίων οργανισμών όπως, όπως η Google και η Amazon που δεν δέχονται τη σωστή αμοιβή των δημιουργών. Πρόκειται για ε, επισφαλή εργασία πλέον των δημιουργών και ε, δίδεται ένα θεσμικό πλαίσιο σε αυτά τα φίλτρα, ενώ υπάρχει συγκέντρωση και μονοπόλιο του ψηφιακού τομέα. Εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε τους δημιουργούς, τους εκδότες, τους συγγραφείς και ούτω καθεξής για να μπορούν να αμείβονται σωστά μέσα στα πλαίσια του εκδημοκρατισμού του πολιτισμού με τη διάδοση περιεχομένου χωρίς ε, φίλτρα και λογοκρισία που ε, προωθούν οι μεγάλες πλατφόρμες που φημώνουν τους δημιουργούς. Η κυρία Βερκούνεν για ένα λεπτό. Arvoisa puhemies, tämä Κυρία Πρόεδρε, η οδηγία δεν είναι τέλεια. Είναι από το κόμμος πέντε των διαπραγματεύσεων και συμβασμών. Ευχαριστώ θερμά τον Άξελ για το έργο του εν μέσω αντιπαρατηθημένων απόψεων. Θεωρώ ότι προστατεύει παρκώ τα δικαιώματα των δημιουργών. Ε, πρόεδρος Ξεκινήστε παρακαλώ από την αρχή λόγω τεχνικού προβλήματος. Κυρία Πρόεδρε, έλεγα ότι η οδηγία δεν είναι τέλεια. Σπάνια έχουμε να κάνουμε τέλεια νομοθετήματα. Είναι από το κόμος πέντε των διαπραγματεύσεων. Συγχαίρω και ευχαριστώ τον Άξελ Φως και όλους όσους συνέβαλαν στο έργο αυτό. Πετύχαμε πολλά. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των δημιουργών και στην ψηφιακή εποχή. Αυτή είναι μια καλή αρχή. Και επίσης, να θυμίσω ότι η οδηγία δεν θίγει την ελευθερία της έκφρασης. Δεν θέτουμε τροχοπέδι σε τίποτα. Έχουμε πλατφόρμες Βεβαίω, εμπορικέ. Εκεί βάζουμε όρια. Και αυτό είναι καλό και για το μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Κέπχατ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγοι για τους οποίους ε, δεν πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτή την οδηγία. Οι νοφείς επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν εξαιρούνται και μετά από τρία χρόνια θα πρέπει ε, να αναλάβουν και να καταστήσουν αυτά τα φίλτρα των μεγάλων επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλο επιχειρηματικό ε, μοντέλο, πολύ επιτυχημένο για τους Αμερικανικούς κολοσσούς. Δεν το θέλουμε όμως, αλλά δεν είμαστε υπέρ της οδηγίας και για κάτι ακόμη, γιατί τελικά δεν φαίνεται να έχει ως στόχο την αναλογική αμοιβή των καλλιτεχνών και δημιουργών. Τα δικαιώματα ιδιοκτησία σε αισθητολογικέ σκέψει έχουν εντελώ αποδυναμωθεί ω προ την ισχύουσα διατύπωση. Αντίθετα, εμεί θέλουμε ισχυρότερα δικαιώματα για του δημιουργού. Αυτά δεν εξασφαλίζονται όμω. αλλά μόνο όσοι εργάζονται ε, σε εκδότε ε, είναι ε, αντικείμενο προστασίας και οι επόμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίε δηλαδή, δεν έχουν αυτή την προστασία και αυτό είναι λάθος. Και κυρία Κώστα, τελευταία ομιλήτρια στο Ευχαριστώ. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, να κατανοήσει ο κόσμος ότι οι δημιουργοί ε, με τη σειρά τους δεν μπορούν να εκμεταλλεύονται και να υποαμείβουν την εργασία των άλλων. Δεν έχει νόημα να υπάρχει εκφοβισμός κατά των Ευρωπαίων πολιτών. Ξέρουμε ότι σήμερα θέλουν να υπερασπιστούν τα εμπορικά τους δικαιώματα. Μην ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη πλατφόρμα έχει ε, υπέρογκα έσοδα από τη διαφήμιση αλλά η Silicon Valley δυστυχώς όπου κι αν βρίσκεται ανά τον κόσμο δεν καταβάλει φόρους. Δεν ήθελα να σας σταματήσω, απλώς να επιβραδύνετε λιγάκι. Έχετε 15 δεύτερα στη διάθεσή σας, αλλά μιλάτε με ταχύτητα φωτός, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα 15 δεύτερα. Δεν σας ακούω, κυρία Κώστα. Έχετε 15 ε, δεύτερα. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι πρόβλημα για μένα. Για μας πρόκειται για μια μεγάλη μάχη για την δημιουργία και τον πλουραλισμό της πληροφορίας. Υπερασπιζόμαστε εκατομμύρια θέσεων εργασίας ε, για τους εκδότες, ε, δημιουργός και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε καταστήλει πολλά fake news, ε, τα οποία θα πρέπει να κατασταλούν. Η Wikipedia πολλές φορές παραπλανά. Κύριε Υπάρχει μια σύγχυση εδώ γιατί δεν σας είχα στον κατάλογό μου. Θα σας δώσω το λόγο. Κύριε Βόρντ, υπάρχουν τόσοι άλλοι που δεν μπορεί να γίνει. Ας ελέγξουμε τις υπηρεσίες πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί ξέρετε το θέμα είναι σημαντικό για τους συναδέλφους. Παρακαλώ κύριε ένα λεπτό αυστηρά. Θα πρέπει να θυμηθούμε γιατί δημιουργήθηκε αυτή η οδηγία. Όχι γιατί υπάρχει δυσκολία πρόσβαση στο ίντερνετ, αλλά επειδή οι πολίτες θέλουν να καρποθούν το αποτέλεσμα της εργασίας τους, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Υπάρχει μεγάλη πειρατεία. Αυτό είναι έγκλημα γιατί δεν υπερασπιζόμαστε τους ε, κανόνες της παραγωγής ε, στην τέχνη, πολιτισμό και δημοσιογραφία αυτό ακριβώς συμβαίνει. Όταν χρησιμοποιούμε μια εικόνα ή ε, ένα συγκεκριμένο έργο ή απόσπασμά του. Εάν ο δημιουργός θέλει να υπερασπιστεί το έργα του, δεν έχει επαρκή μέσα για να το κάνει στον ψηφιακό χώρο. Είναι όνειδος αυτό, το ότι δεν δίνουμε τη δυνατότητα αυτή στους δημιουργούς. Γκραπίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε. Καθίσταται σαφές ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τομέα τον οποίο θα πρέπει να ρυθμίσουμε. Όλα ξεκίνησαν από την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία του εκφράζεστε, αλλά και προστασία του δημιουργού και ανταμοιβή της εργασίας. Χρειαζόμαστε όμως και μία δημιουργική βιομηχανία. Δεν μπορούμε χωρίς πολιτισμό. Βεβαίως τα άρθρα 11, 13 και 14 είναι χρήσιμα. Όλοι συζητήσαμε με όλους και θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτά τα άρθρα για να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός και να βελτιώσουμε αυτή την οδηγία. Αν δεν κάνουμε όμως τίποτα, δεν νομίζω ότι η ψηφική αγορά θα προστατευτεί περισσότερο. Δεν θα ε, προστατεύσουμε τους δημιουργούς. Τα άρθρα αυτά έχουν έχουν αλλάξει. Καπούτο ένα λεπτά. Ξέρω ότι μερικοί είναι δυσαρεστημένοι που δεν θα τους δώσω το λόγο. Καπούτο. Είναι τρίτη φορά που παρεμβαίνω για την οδηγία copyright. Στην αρχή μίλησα για αναπομπή στην Επιτροπή για καλύτερη εξισορρόπηση, ιδιαίτερα στην περίπτωση αναπαραγωγής. Η οδηγία για την πνευματική οδιοκτησία θα βοηθήσει στην ανταμοιβή των δημιουργών. Αυτή τη στιγμή δέχομαι χιλιάδες mail από διάφορα λόμπι για να ε, συνεχίσουν τα προνόμια που είχαν κατά το, τα πρώτα χρόνια του 2000, την πρώτη δεκαετία δηλαδή ε, και γι' αυτό δεν νομίζω ο, παρά να λάβουμε υπόψη τους τριμερείς όπου απαγορεύεται η λογοκρισία και υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο διαδίκτυο και για όλες τις πλατφόρμες. Η κυρία Γουιλάρ Γκαρθία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η συζήτηση και αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι πολύ ε, αμφιλεγόμενη και επίμαχη. Όχι γιατί υπάρχει αποκλήση απόψεων, κάτι που είναι καλό σε κάθε συζήτηση, ήθιστε να υπάρχουν αποκλήσει απόψεων, αλλά είναι πολύ περίεργο. Μιλάμε για έναν απαραίτητο κανονισμό που θα ρυθμίσει την ψηφιακή αγορά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλο πάθος. Ε, εμένα κάπως με ξενίζει, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στρέβλωση στην ενιαψηφιακή αγορά και με τον κανονισμό, με την οδηγία μάλλον αυτή, ο στόχος είναι ε, προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού και νομίζω ότι είναι ισορροπημένη πρόταση. Γιατί είμαστε λοιπόν αντίθετοι σε αυτή τη ρύθμιση. Η ρύθμιση δεν σημαίνει απαγόρευση. Απλά σημαίνει ότι μπαίνουν κανόνες, έτσι ώστε όλοι σε αυτήν την αγορά και στη ψηφιακή αγορά ε, και στην εμπορική και τη χρηματοπιστωτική αγορά να γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Μόνο περί αυτού πρόκειται. Πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε υπέρ ε, της οδηγίας αυτής. Ευχαριστώ. Κυρία Ward. Ως εκπρόσωπος των εργατικών για τον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι πρέπει να υπερμηνθούμε των μικρομεσαίων που εργάζονται στο δημιουργικό. Πρόκειται εδώ για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση εδώ και 15 χρόνια και θα σταματήσει επίση του γίγαντε από τι επεμβάσει του στο διαδίκτυο. Ακόμη πιο σημαντικό, διασφαλίζει η οδηγία, ότι οι δημιουργοί απολάβουν αξιοπρεπού αμοιβή. Αυτό το πακέτο μεταρρύθμιση κάνει κάτι επιτέλου για την σημερινή κατάσταση όπου ένα τραγούδι μπορεί να, να μεταδοθεί 50 εκατομμύρια φορές πριν ε, ο δημιουργός του μπορέσει να διεκδικήσει κάποια αμοιβή. Αυτό θέλουμε, να αναγνωριστούν και να μειφθούν επαρκώς οι δημιουργοί. Η, δημιουργία, η οδηγία αυτό κάνει, αποτελεί επένδυση στον τομέα του δημιουργικού. Θέλω να ευχαριστήσω τις ενώσεις των καλλιτεχνών στο Ηνωμένο Βασίλειο Διακόπτη πρόεδρο. Πρέπει να σα διακόψω και τώρα ο επίτροπο Ανσίπ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συζήτηση. Πολλοί μιλητές αναφέρθηκαν στο φίλτρο, στο περίφημο φίλτρο το οποίο δεν αναφέρεται όμως στο κείμενο της οδηγίας. Όπως γνωρίζουμε, χρησιμοποιείται από τις μεγάλες πλατφόρμες. Η καταψήφιση της οδηγίας δεν θα καταργήσει τα φίλτρα αυτά. Η οδηγία των αντίων θα δώσει στους πολίτες μας το δικαίωμα να ζητήσουν την αφαίρεση υλικού για το οποίο πρέπει να λάβουν αμοιβή. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Η ψηφοφορία αφορά το μήνυμα που θέλει να στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δημιουργούς της. Και είναι απλά τα πράγματα. Φροντίζουμε για σας, σας έχουμε στο μυαλό μας και σας προστατεύουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, για να μπορέσετε να συνεχίσετε το πολύτιμο έργο σας και να συμβάλλετε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι θεμέλιο της κοινωνίας μας. Είναι πηγή των αξιών μας και της έμπνευσής μας. Η τελική δικαιούχοι, αν θέλετε, αυτής της οδηγίας είναι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σύγχρονο περιβάλλον για τα πνευματικά δικαιώματα σημαίνει πρόσβαση στην ψυχαγωγία, στην δημοσιογραφία και Γι' αυτό το λόγο η ψηφοφορία αφορά τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζει τις πολύπλοκες νομικές προκλήσεις του διαδικτυακού περιβάλλοντος. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διστάμενες απόψεις και αυτό είναι καλοδεχούμενο στο πλαίσιο ενός διαλόγου. Αφού γραστήκαμε τις διστάμενες απόψεις, δείχνουμε σεβασμό όμως πιστεύουμε ότι εν τέλει το κείμενο από το του τριμερούς διαλόγου είναι ισόρροπο και επιτελεί ακριβώς τον στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή, τον εξυγχρονισμό του δικαίου μας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να ετοιμαστούμε για την ψηφιακή εποχή. Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τους και οδησίες ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Άνσιπ. Καλωσορίζω όλους και πάλι. Συνέχιζω να προεδρεύω κύριο Φως. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε στη σημερινή συζήτηση ε, και από κάποιες παρεμβάσεις ε, ξαναβλέπουμε ότι κάπως έχασε το μέτρο αυτή η συζήτηση. Δεν θα υπάρξει λογοκρισία με αυτή τη μεταρρύθμιση η ε, ελευθερία έκφραση, η νόμιμη, δεν θα περιοριστεί με αυτή την έκθεση. Εμείς καταφέρνουμε να έχουμε ε, ασφάλεια δικαίου ε, και νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, οι χρήστες, οι πολίτες έχουν περισσότερα δικαιώματα και ελευθερία, Facebook, Google, YouTube κτλ. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν παραπληροφορούν και βάζουν πάρα πολλά λεφτά για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και δείχνουν πόσο εύκολο τελικά είναι ε, τις ε, ομάδες των νέων, την νεολαία, να τις ε, χειραγωγήσουν και να τις επηρεάσουν. Σήμερα το Κοινοβούλιο, η Δημοκρατία μας δεν στρέφεται κατά τον, και δεν θέλει να επιβληθεί σε βάρος των κολοσσών του διαδικτύου, αλλά να εξασφαλίσει την προστασία ε, της πνευματικής δεξίας, γιατί γι' αυτό μιλάμε, για την πνευματική δεξία, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, θέλουμε δίκαιη αμοιβή των δημιουργών. Αυτή είναι η στόχη μας και είναι στο δικό μας χέρι σήμερα να σώσουμε ε, την ευρωπαϊκή πολιτιστική δημιουργία. Δεν θέλουμε εκμετάλλευση από τα μονοπόλια. Ε, στο χέρι μας είναι σήμερα να προσφέρουμε την ε, απαραίτητη και την αναγκαία προστασία ε, στους ε, κλάδους της δημιουργικής πολιτιστικής βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φως, λέει ο Πρόεδρος. Εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε και σήμερα για την έκθεση αυτή. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, ε, την έκθεση του κυρίου Κοτσολίνο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Ταμείο Συνοχή. Καταρχά, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Κοτσολίνο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα ψηφίσουμε και θα δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ισορροπημένο ε, κείμενο. Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Σύνοχης είναι τα μεγαλύτερα μέσα χρηματοδότησης για την επταετία 21-27. Και θεωρούμε ότι παρόλα αυτά υπάρχουν ε, στοιχεία που δεν μπορούμε να ε, δεχτούμε. Δεν μπορεί να υπάρχει ε, διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καλύτερη ποιότητα ζωής όλων των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες. Αυτό είναι ένα μέσον για να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, να εργαστούμε για να μην μείνει κανείς πίσω. Καμία περιφέρεια, ούτε η εξόχως απομακρυσμένες. Αυτό ίσχυε για την Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία, καθώς και την Ιταλία μετά από τους σεισμούς. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα πολιτιστικά αγαθά, τα οποία πολλές φορές ε, καταστρέφονται. Η πολιτική λιτότητας οδήγησε σε μια δραματική μείωση πόρων και γι' αυτό η περιφερειακή πολιτική αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία και γι' αυτό οι δημόσιες επενδύσεις δεν μπορούν να περιοριστούν στο ίμιση. Πέντε είναι οι προτεραιότητες στο νέο κανονισμό. Καινοτόμα και ευφύς ανάπτυξη. Μια Ευρώπη πιο πράσινη με μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για να προωθήσουμε την ενεργειακή μετάβαση, μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη και πιο κοινωνική, χωρίς αποκλεισμούς, για μια νέα ευημερία των πολιτών και μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες ε, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς των εξόχως απομακρυσμένων περιοχών. Αυτή είναι η πολιτική συνοχής. Έχουμε μια συγκεκριμένη θεματική έτσι ώστε για όλες τις περιφέρειες να ε, προσδώσουμε το 30% των πόρων. Επίσης υπάρχουν στοιχεία ευελιξίας έτσι ώστε να προωθήσουμε την τοπική ανάπτυξη. Μιλάμε για ένα 10% προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και ένα 5% το οποίο προορίζεται στις μικρές κοινότητες, τις απομακρυσμένες, τις ορεινές περιοχές. Επίσης μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημόσια διοίκηση και έχουμε και μέσα ευελιξίας για συγχρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ καλή αυτή η εργασία και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συνεισέφεραν τώρα. Εμείς θα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε στο σώμα αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, ιδιαίτερα ως προς το κλιματικό και τα περιβαλλοντικά. Αλλά ας είμαστε σύσσωμοι στην ε, ψηφοφορία έτσι ώστε το επόμενο κοινοβούλιο να έχει ένα συνεκτικό μέσο υπεράσπισης του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής. Η κυρία Βέρα Γιούροβα έχει το λόγο, η Επίτροπος. Η ψηφορία αύριο είναι σταθμός στην επιμερισμένη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Ταμείων και το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Τα δύο βασικά εργαλεία επενδύσεων στην ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος και τις υποδομές. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κοτσολίνο, τον εισηγητή, καθώς και τους άλλους βουλευτέ, μέλη τη Επιτροπή ε, Περιφερειακή Ανάπτυξη, αλλά και στι άλλε επιτροπέ για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του έργου του υπό μεγάλη χρονική πίεση. Λυπούμε μόνο που οι εκλογέ του Μαΐου είναι πολύ κοντά. Και ω εκ τούτου, βρισκόμενοι ακόμη στην πρώτη ανάγνωση, θα επιτρέψει ε, την συνέχιση αυτού του έργου κατά τη διάρκεια της παρουσιαστητίας. Αν διαβάσει κανεί την έκθεση της Επιτροπής ε, Ρέτζι, το Κοινοβούλιο αξιολογεί θετικά τι περιφερειακέ παρεμβάσεις σε όλη την Ευρώπη, ώστε να μην μείνει πίσω καμία περιφέρεια. Εν τούτης, παρά το ότι συμφωνούμε με τους στόχου, δεν συμφωνούμε πάντοτε με τα εργαλεία, με τα μέσα. Και επιτρέψτε με εδώ να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Η θεματική συγκέντρωση και το πεδίο εφαρμογή της υποστήριξης. Επικεντρωνόμαστε σε ολιγάριθμες πρωτοβουλίε. Θεμερικέ πρωτοβουλίε. και αυτό είναι καλό για την αποτελεσματικότητα των δαπανών μας. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή την θεματική στόχευση χωρίς να ξεχνούμε τους βασικούς μας στόχους, την ευφιέστερη και πιο καθαρή Ευρώπη. Να ασχοληθούμε με το περιβάλλον και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό όμω δεν σημαίνει περισσότερη συγκέντρωση. Αντιθέτω, θα είμαστε πιο ευέλικτοι στην υλοποίηση των πακέτων. Όσον αφορά τις περιφέρειες, πιστεύω ότι μπορούν να συμμετάσχουν και με δικούς τους πόρους. Όσον αφορά τώρα τα τρία επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό, μπορούμε να πετύχουμε συνέργεια εύκολα. Και όσον αφορά τους στόχους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σαφέ όραμα μιας πιο κοινωνικής και καλύτερα διασυνδεμένης Ευρώπης. Όσον αφορά τους, επιπλε, τους επιμέρους στόχους, το δεύτερο επίπεδο, αυτοί δεν αναφέρονται εξαντλητικά βεβαίως, όσον αφορά τι επιλέξιμε ε, δράσει. Διατυπώνουμε γενικού στόχου εδώ. Και αυτό ήταν άλλο ένα βήμα. Περάσαμε ε, από τον προσανατολισμό στις δράσεις στον προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Ευτυχώ από ε, αυτού καταφέραμε να πετύχουμε συνεννόηση. Επαναπροσδιορίζουμε λοιπόν τους στόχους. Όπως είπε και το Κοινοβούλιο και ιδίω όσον αφορά την κινητικότητα στις πόλεις, τους φυσικούς ε, πόρους, ε, τη διασυνδεσιμότητα κλπ. Έτσι, παρά τους θεματικούς στόχους, ενθαρρύνουμε ευρύτερες επενδύσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις τοπικές ανάγκες. Επίσης, αποκλείσαμε, πες προτασιός μας, Κάποιου θεμετικούς στόχους που θεωρούμε ότι έχουν χαμηλέ θετικές επιπτώσεις. Ας πούμε, επενδύσεις σε χώρου υγειονομική ταφή ή σε δράσεις που μας δεσμεύουν για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, επενδύσει στα ορυκτά καύσιμα. Φοβούμεθα ότι κάποιε τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα βοηθήσουν. Όμως η Κομισιόν θέλει να τονίσει ότι οι διατάξεις που αφορούν το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας δεν είναι καλό να εφαρμοστούν μέσω τομεακής νομοθεσίας. Προτείναμε αντιθέτω ο κανονισμός κοινών, κοινών διατάξεων να διέπεται από την αρχή της, των μακροοικονομικών ε, προϋποθέσεων. Προσβλέπω σε μια επικοδομητική συζήτηση. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Κυρίε και κύριοι, λέει ο Έχουμε την Επιτροπή Προπολογισμών, ε, Ελέγχου του Προπολογισμού, ε, Περιβάλλοντο, Τραν, την Άγκρη και την Επιτροπή Πολιτισμού που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα. Οπότε ξεκινούμε τη συζήτηση εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Πρώτα όμω η Επιτροπή Προπολογισμών, ο κ. Ολμπρέχτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ακούσαμε με ενδιαφέρον τα όσα είπατε, καθώς και τα κριτικά ε, σχόλια που εκφράσατε για τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, να ξεκινάει έτσι η συζήτηση. Είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα το Κοινοβούλιο. Στήριξε την Κομισιόν σε ό,τι αφορά την απλούστευση της δικασίας ε, και συμφωνούμε με ορισμένου από του στόχου σα, δηλαδή για ε, σαφήνεια, διαφάνεια των στόχων για τις αστικές μεταφορέ. Όμω, το Κοινοβούλιο έχει αποκλίνει σε ορισμένα σημεία από το κοινοβούλιο, από την Επιτροπή σε τέφερα κάποιους ομονωμένου στόχους, όχι γιατί θέλουμε λιγότερη αποτελεσματικότητα, αλλά περισσότερη συνοχή. Εξού και έχουμε κάπως ε, διαφοροποιηθεί για τον αποκλεισμό ρημένων ομάδων, τις θελματικές πλατφόρμες και τις επενδύσεις. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά, ε, είναι μια καλή πρόταση. Όμως, κατά την άποψη του Κοινοβουλίου, γι' αυτό απαιτούνται αλλαγέ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Μέρος Επιτροπή Έλεγχου του Περιπολογισμού, κ. Ντέρεκ Βον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Το ΕΤΠΑ θα παραμείνει ένα βασικό επενδυτικό εργαλείο για την Ένωση για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθότι θα ανέρχεται περίπου στο 25% του προϋπολογισμού. Επιτροπή Ελεκτού του Προϋπολογισμού σίγουρα ε, θα εξασφαλίσει τη σωστή ε, αποτελεσματική διαχείριση και δαπάνη των ελόγων κονδυλίων. Αναγνωρίζουμε όμως ότι το Ταμείο είναι σημαντικό ε, και εξού καλωσορίζουμε τις περισσότερες από τις προτάσεις του εισηγητή. Αντίθετα ίσως από την Κομισιόν. Θέλω ιδιαίτερα να επικροτήσω ρωτήσω την πρόταση ε, να δοθούν κάποια κονδύλια για πρώτη φορά στην Ήπετρο σε αγροτικέ περιοχέ. Γιατί κάτι των παρελθόν ξέρουμε ότι ένιωσαν ότι ε, είναι κάπως παραγνωρισμένες αυτές οι περιοχές στο πλαίσιο του Τόμιου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. Ε, ίσως ε, η Ουαλία να μην ωφελείται στο μέλλον από τα κονδύλια συνοχής ε, παρότι μέχρι τώρα ωφεληθήκαμε τα μάλα. Παρ' όλα αυτά μεγάλη χρηματοδότηση παρέχει το ΕΤΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει εντό Ένωση και να συνεχίσει να ωφελείται από το Ταμείο αυτό. Εμεί θα συνεχίσουμε πάντω να αγωνιζόμαστε υπέρ αυτού του Ταμείου και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος εκ μέρου τη Επιτροπή περιβάλλοντο Το λόγο έχει η κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπα, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα σας μιλήσω εκ μέρους της δικής μου επιτροπής και θα εκφράσω την άποψή μας. Εμείς συμφωνούμε ότι περισσότεροι πόροι πρέπει να διατεθούν για τη βελτίωση των αποδομών στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούν να, να ε, εκπληρώνουν τους στόχους για τις μεταφορές, για τα απορρίμματα και απόβλητα, για την αλλαγή του κλίματος. Ε, το Ταμείο Συνεχής είναι ένα πολύ σημαντικό ταμείο οι πόροι ε, του Ταμείου Συνοχή μπορεί να είναι και το 50% των δημόσιων επενδύσεων για κάποιε χώρε. Χωρί αυτά τα κονδύλια δεν θα μπορέσουν οι χώρε αυτέ να προβούν σε εξυγχρονισμό. Είμαι απογοητευμένη που η Επιτροπή Ρέγγι δεν σεβάστηκε τι αποφάσει τη Επιτροπή ΕΝΒΗ ε, για την πολυτροπικότητα και του στόχου τη κινητικότητα. Να πάνε από τον στόχο 3 στο στόχο 2. Θέλουμε να έχουμε λιγότερες εκπομπές από τις μεταφορές για να γίνουν σεβαστοί στόχοι του κλίματος. Άρα περισσότερα κονδύλια πρέπει να διατεθούν για την πρόθεση των ε, οχημάτων που εκπέμπουν ε, λίγα καυσαέρια. Πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος Επιτροπής Μεταφορών, η κυρία Ρεόντα Λον Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η αναθεώρηση αυτών των ταμείων είναι μείζωνος σημασίας για τις περιφέρειες. Για να γίνει χρηματοδότηση των περιφερειών θα πρέπει να γίνει χρηστή διαχείριση πολύ πιο κοντά στους πολίτες και να υπάρχει και ένα περιθώριο ελιγμού στις τοπικές αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. ω εισηγήτρια από την Επιτροπή Μεταφορών θα ήθελα να σταθώ στην ιδέα της Επιτροπής που προβλέπουν αποκλεισμό των σιδηροδρόμων και των αεροδρομίων από αυτό το πλαίσιο. Νομίζω όμως ότι για να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη και σωστή ανάπτυξη θα πρέπει οι περιφέρειες να μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές μεταφοράς όπως επιθυμούν, ως προς τα αεροδρόμια που αποτέλεσαν αντικείμενο ζωηρών συζητήσεων εδώ, η πολιτική μου οικογένεια υπέβαλε τροπολογίες για τα παλαιά αεροδρόμια έτσι ώστε να υπάρχει αναβάθμιση του περιβάλλοντος και για να ε, καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Έχετε υπερβεί το χρόνο σας. Θα είμαι πολύ αυστηρός διότι έχουμε πάνω από 10 λεπτά καθυστέρηση και θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 12.30. Εξ ονόματος της Επιτροπής ε, Γεωργίας, ο κύριος Νίκολσον, ο οποίος δεν είναι παρόν, άρα ο κύριος Ντρογεύσκη έχει το λόγο. Πρόεδρε, να σας υπενθυμίσω κάτι. Πάμε πίσω στις αρχές αυτής της θητείας. Δεν θα πω ότι η πολιτική συνοχής ε, δέχονταν επικρίσεις, αλλά υπήρχαν Εγώ Τότε ήμουν υπουργό πολιτισμού και στην Πολωνία Εν μεταξύ, καταφέρουμε να κάνουμε πολλά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Πολλοί μαζιλεύουν για αυτά τα οποία κατορθώσαμε χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Σήμερα η πολιτική συνοχής είναι εμπεδομένη, ευρέως αποδεκτή, θεωρείται σημαντική, απολάβει σεβασμού και γι' αυτό την χρηματοδοτούμε ακόμη περισσότερο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Όλμπρεχτ και την κυρία Χούμπνερ που υπερψήφισαν και υπόθεσαν μάχη για την πολιτική συνοχή. Είναι μια πολιτική που πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω. Βεβαίω προ τούτο πρέπει να θέσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένου στόχους για να αποκρούσουμε και τι άτοπε επικρίσεις. Σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων, όμω γενικά το κείμενο είναι εξαιρετικό. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Πολιτικές ομάδες. Λουίς Βαλκάρτελ Σίσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αύριο θα ψηφίσουμε σε πρώτη ανάγνωση τη θέση μας για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Νομίζω ότι χάρη στην εργασία των τελευταίων μηνών καταφέραμε να βελτιώσουμε την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Θα θέλαμε το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής να χρηματοδοτήσουν τις έκτακτες ε, καταστροφές όπως σεισμούς, πλημμύρες κλπ. Ε, για να μην φτάσουν τα χρήματα αργά για την αντιμετώπιση μιας φυσικής ε, καταστροφής. Εδώ θα πρέπει να δούμε και τις εξόχως απομακρυσμένες ε, περιοχές και να δούμε και το πρόβλημα του αποπληθισμού και το θέμα των, των μικρών θυλάκων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα ήθελα να πω ότι χάρη στη κοινή εργασία μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της απομάκρυσης του πληθυσμού από ορισμένε περιφέρειες, ιδιαίτερα σε σχέση με την πράσινη οικονομία και την κοινωνική καινοτομία. Να μπούμε σε μία δημογραφική άνοιξη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε, να δώσουμε εγγυήσει σε αυτούς που θέλουν να προωθήσουν μία βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό αφορά τα ψηφιακά της δημόσιες υπηρεσίες και τα βοηθήματα για τη μητρότητα. Εάν μιλάμε για μία αγροτική Ευρώπη θα πρέπει να κάνουμε πολλά ε, φτάσαμε στην ολοκλήρωση ενός συστήματος με βάση τις κοινέ ευκαιρίες και τα κοινά προστάγματα που υπάρχουν για τις οικογένειες και τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Έχουμε και πολλούς ε, ε, συμμετέχοντες στα, στα ε, θεωρία Μποστινάρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοτσόλου. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία και ο ίδιο εργάστηκε πολύ καλά. Εγώ έχω διατελέσει και για το Ταμείο Σύνοχη κατά το παρελθόν. Δεν είμαι ικανοποιημένη.